Okay, the problem is solved. Ωραία λύθηκε το πρόβλημα. Οπότε... Να δώσω το λόγο στο συντάκτη μιας μελέτης που αφορά αυτές τις επιχειρήσεις. Καθηγητής Φίτση από το Πανεπιστήμιο του Μολύσε. Δέκα λεπτά κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Από τη συνάδελφη. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω καταρχάς ως Κοινοβούλιο και Κομισιόν για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω αυτό το θέμα της κοινωνικής οικονομίας με το οποίο έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια. Τα κυριότερα θέματα που με απασχόλησαν παρόλο που εδώ βέβαια δεν μπορώ να καλύψω όλα τα σημεία που καλύπτει η έκθεση, που είναι λεπτομερής, θα καλύψω μόνο τρία κυρία ζητήματα. που αφορούν ένα ευρωπαίο καθεστώ κοινωνική επιχείρηση. Να δούμε καταρχά αν υπάρχει ευκαιρία ή σκοπιμότητα για ένα τέτοιο καθεστώς και κατά πόσο αυτό ωφελεί την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα και τους πολίτες μας. Βεβαίω, το πρώτο ερώτημα το παντάμε θετικά. Και το δεύτερο είναι τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, τι χαρακτηριστικά έχει. Και τρίτο, αν αυτό το καθεστώς ευρωπαϊκής επιχείρησης, κοινωνικής δηλαδή, είναι κάτι το εφαρμοστέο ή αν παραμένει σε γενικό επίπεδο και αόριστο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να διερευνήσουμε τους πιθανούς τρόπους υλοποίησης αυτού του πιθανού καθεστώτος επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την εταιρική νομοθεσία, το εταιρικό δίκαιο και τη μορφή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα κυρία λοιπόν ζητήματα που διερευνώνται στην μελέτη, μεταξύ άλλων βεβαίως, που δεν θα καλύψω εδώ. Για το πρώτο ζήτημα, κατά πόσο είναι απαραίτητο ή σκόπιμο για την ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων να υπάρχει συγκεκριμένο δίκαιο και καθεστώς για αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα και η απάντηση της έκθεσης είναι καταθατική. Και εξαρτάται από τα προφίλ που αναφέρει η έκθεση. Η σημασία αυτού του ευρωπαϊκού Καθεστώτο κοινωνική επιχειρηματικότητα ε, επιχειρηματικότητας αναφέρεται στα έγγραφα διαφόρων θεσμικών οργάνων. Πολλές χώρες ήδη έχουν κάποιο εταιρικό δίκαιο που αφορά αυτής της επιχειρήσης κοινωνικής ευθύνης. Και θα δείτε τους κύριους λόγους οι οποίοι είναι προφανείς. Δηλαδή, αυτό καθεστώς θα βοηθήσει την ανάπτυξή τους στην Ευρώπη. Θα μπορούσε επίσης αυτό ο καθεστώς επιχείρησης κοινωνικής επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικότητας θα μπορούσε λοιπόν να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες αυτής της μορφής επιχειρηματικότητας. Βεβαίως, μαζί με ένα ισχυρό δημόσιο νομικό πλαίσιο που θα αφορά αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις και το οποίο σε κάποιες χώρες ήδη υπάρχει. θα επιτρέψει βεβαίως και στις επιχειρήσεις αυτές να μην μεταβάλουν τη φύση τους και να τη διατηρήσουν. Επίση, θα μπορούσε να μα βοηθήσει στο να μπορούν να συμμετάσχουν αυτές οι επιχειρήσεις και σε διάφορες νομικές διαδικασίε που αφορούν και τις υπόλοιπε επιχειρήσεις, α πούμε σε διαγωνισμούς, δημόσιες προμήθειε κλπ. ώστε να αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο η ορατότητα, η παρουσία των επιχειρήσεων αυτών των κοινωνικών. Έχουμε επίσης και το θέμα της κοινωνική ευθύνη. Η κοινωνική ευθύνη, όπως έχουν επαγγελμένως πει τα ευρωπαϊκά όργανα, είναι κάτι το οποίο αφορά τις κανονικές επιχειρήσεις και έχει σχέση με τις κοινωνικές τους δράσεις. Ενώ για τις κοινωνικές επιχειρήσεις η προϋπόθεση είναι ακριβώς να επιχειρούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε στην ομοθεσία μας αυτή τη διάκριση. Και μιας και μιλάμε για διάκριση, για διευκρίνηση, υπάρχει μια παράγραφο στην έκθεση που παρουσιάζει ακριβώς τη διαφορά μεταξύ κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως συγκεκριμένου φορέα της κοινωνικής οικονομίας και της έννοιας της κοινωνικής ευρύτερης οικονομίας που περιλαμβάνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα αλλά πηγαίνει και παραπέρα Πρέπει λοιπόν να κάνουμε όπως έλεγε, αυτή τη διάκριση. Ένα άλλο θέμα, αφού ρυθμίσουμε το πρώτο που ανέφερα, λέγοντα ότι ναι, θα ήταν πολύ καλό να έχουμε ένα ευρωπαϊκό καθεστώ κοινωνική επιχείρηση. Ένα δεύτερο θέμα που σχετίζεται εδώ είναι το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά αυτού του ευρωπαϊκού καθεστώτος. Στην έκθεση μελετάμε 18 εθνικά καθεστώτα κοινωνικής επιχείρησης και προσπαθώ να τα ταξινομήσω τα καθεστώτα αυτά σε κάποιες κατηγορίες. Οι κύριες διαφορές που βρήκα και που θα πρέπει να λάβει υπόψη ο Ευρωπαίος νομοθέτης είναι αυτής είναι αυτή που αφορά κάποια συγκεκριμένη μορφή κοινωνική επιχειρηματικότητα όπω κοινωνικό συνεταιρισμό που έχουμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και σε άλλε χώρε τη Ένωση και εκτό Ένωση και κοινωνική επιχείρηση ω νομικό χαρακτηριστικό ιδιότητα. Αυτό είναι σημείο κλειδί για την νομοθεσία, για να κατανοήσουμε ακριβώ τη φύση τη κοινωνική επιχειρηματικότητα. Όταν κοινωνική επιχείρηση είναι συγκεκριμένο είδου ή υποείδου, νομικού, νομικής οντότητας, τότε μπορεί να έχουμε μορφή εξεντεριστική ή κοινωνική. Ενέδωση, δηλαδή κοινωνικής επιχείρησης όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που ασκούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα κοινωνική που δεν γίνεται κερδοσκοπικά αλλά προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Όταν λοιπόν υιοθετούμε, υιοθετήσουμε αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να επιλέξουμε και τη νομική μορφή της κοινωνικής επιχείρησης, αυτή που θα πρέπει να έχει κοινωνική επιχείρηση. Στο δεύτερο πρότυπο της νομοθεσίας, θα πρέπει να δούμε τις νομικές κατηγορίες, ομάδες και καθεστώτα επιχειρήσεων. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να το κάνουμε βάσει της νομικής μορφής της κοινωνικής επιχείρησης. Το οποίο σημαίνει ότι η κοινωνική επιχείρηση θα μπορούσε να συσταθεί υπό διαφορετικέ νομικέ μορφέ. Μέσω συνεταιριστική μορφή, ε, συνεργατική, οτιδήποτε. Έχουμε λοιπόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία θα αναλύσω στη συνέχεια. Και μετά βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν θα εξηγήσω εδώ. Αλλά τους παρουσιάζω στην έκθεση. για συγκεκριμένες κατηγορίες κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες θα ήταν προτιμητές σε περίπτωση που νομοθετήσουμε για αυτές τις επιχειρήσεις και που ανταποκρίνονται σε πρακτικές που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο οι εθνικοί νομοθέτες. Γιατί έχουμε την τάση όλο και περισσότερο στην Ευρώπη να έχουμε ένα καθεστώς κοινωνικής επιχείρησης και αυτό να καλύπτει διάφορες επιχειρήσεις που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Η άλλη διάκριση είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις κοινωνικής ολοκλήρωσης. Είναι επιχειρήσεις που ασκούν διάφορες δραστηριότητε κυρίως υπέρ ατόμων μειονεκτούντων, οπότε θα ήταν καλύτερο κατά την άποψή μου να μην περιοριστούμε στο στοιχείο της εργασίας ένταξης δηλαδή στην εργασία το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα χαρακτηριστικό αλλά όχι αποκλειστικό όσον αφορά την νομοθεσία που θα διέπει αυτέ τι κοινωνικέ επιχειρήσει. Τελευταίο σημείο σε αυτή τη διαφάνεια για τα μοντέλα που θα εθετήσουμε ανεξάρτητα επιλογή θα πρέπει να ποια είναι τα χαρακτηριστικά τη κοινωνική επιχείρηση. Απαριθμούνται αυτά είναι ιδιωτικέ επιχειρήσει ανεξαρτήτω ή εκτό κράτου, οι οποίε διαδραματίζουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή έχουμε μια εταιρεία μη κερδοσκοπική, αλλά προ το συμφέρον, προς το καλό του κοινωνικού συνόλου. Σύμφωνα με μια κοινωνική υπηρεσία, συμμετοχή κοινωνικών φορέων και ενίσχυση και του κοινού, του κοινωνικού συνόλου. Να πω εδώ ότι αν δούμε το καθεστώς αναρμόνισης του, κοινωνικού, του εταιρικού δικαίου στην Ευρώπη, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Και αν δούμε και τις υπερεθνικές νομικές μορφές των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, τα πράγματα είναι λίγο απογοητευτικά, γιατί ξέρετε ότι η εργασία για αυτές τις επιχειρήσεις, τις συνεργατικές και άλλες, έχει σταματήσει. Γι' αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αρνητική στάση προ μια ενδεχόμενη εναρμόνιση εκ μέρου τη ΕΕ στι χώρε μέλη. Εγώ προτείνω να διερευνήσουμε το εξή στο εταιρικό δίκαιο. Να υπάρχει ένα είδος μονοπρόσωπης επιχείρησης το οποίο το προτείνω ως ενδεχόμενη λύση για το πιθανό καθεστώς κοινωνική επιχείρησης. Αυτά συμπεράσματα Ξαναλέω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα καθεστώς κοινωνική επιχείρησης, αυτό το συμπέρασμα της δουλειά μας, και να εργαστούμε όχι μόνο στις κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά ευρύτερα σε όλες τις φάσεις κοινωνικής οικονομίας, και των επιχειρήσεων που δεν περιορίζονται μόνο στις κοινωνικές επιχειρήσεις και πρέπει να πούμε ότι είναι επίσης σημαντικό να ολοκληρώσουμε το πλαίσιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα που θα, θα εμπλέξει, θα περιλάβει όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας αυτού του είδους. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγήτα. Και τώρα ο καθηγητής Μερσλάιν, καθηγητής uh, business στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ. Και καθηγητά έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι κάτι που έχει διαφορετικές πτυχές. Βιομηχανία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί που ξεκινάνε από τα αυτοκίνητα μέχρι και παγωτά Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις δεν είναι οι παραδοσιακές, δεν είναι φιλανθρωπικές, είναι οικονομικές, ε, οι οποίες παράγουν σε τιμές της αγοράς. Και το μόνο που λείπει είναι να υπάρχει κάποια κοινωνική ευθύνη. Ε, δυστυχώς, ε, μάλλον για να το πω αλλιώς, ότι ε, όσον αφορά τις ε, παραγωγές ε, για τις οποίες μιλάμε, αυτές έχουν ως κύριο στόχο το κέρδος. Και οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν και το κέρδος με την κοινωνική συμπεριφορά, την επιχειρηματικότητα. Διακόπτει ο πρόεδρος. Αν έχει την καλοσύνη να μιλάτε πιο αργά, λέει ο πρόεδρος διακόπτοντας τον ομιλητή. Υπάρχει και ένας τέταρτος τομέας παράλληλα με τις ιδιωτικές ε, και τις κοινοφελείς επιχειρήσεις, ένας τομέας ο οποίος ε, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Για μας τους νομικούς ε, και για εσάς που είστε ειδικοί επί των νομικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον για αυτόν τον τομέα είναι να υπάρχουν νομικοί κανόνες, κατά πόσον δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή στο εταιρικό δίκαιο. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον οι υπάρχουσες δομές ε, δεν μπορούν να συνδυάσουν το κοινωνικό στοιχείο με το στοιχείο του κέρδους. Δηλαδή ε, είτε θα πρέπει να ισχύει το ένα είτε το άλλο. Στις κεφαλογικές εταιρείες ε, και στις μετοχικές εταιρείες υπάρχει το στοιχείο του μετόχου. Η διοίκηση είναι, να, είναι αναγκασμένη να καταβάλει μερίσματα ο περιορισμός είναι ο ε, σημαντικότερος λόγος γιατί οι ΗΠΑ ε, έχουν εισαχθεί νέες μορφές εταιριών. Ε, σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η διοίκηση έχει περισσότερο περιθώριο αλλά πολλές φορές είναι ασαφή τα όρια. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πολλές εταιρείες δεν αναπτύσσουν κοινωνική δραστηριότητα. Σε κάποιο εταιρικό δίκαιο υπάρχει και κάποιο περιθώριο για τους μετόχους, όπως το καταστατικό αναφέρεται ότι η εταιρεία ε, μπορεί και θέλει να ε, λειτουργεί ε, κοινωνικά. Στην Γερμανία υπάρχουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί. Επίση, αυτό που είναι προβληματικό είναι ότι αλλάζει κάθε τρεις και λίγο το κατσατικό, παρήματος χάρη ε, όταν ε, εξαγοράζεται η εταιρεία. Εκτό αυτού υπάρχουν και άλλοι λόγοι γιατί πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώ. Δηλαδή οι εταιρείε ε, οι οποίε τάσσονται υπέρ ενό τέτοιου ειδικού καθεστώτο, οι εταιρείε αυτέ μπορούν να δώσουν ένα μήνυμα ότι λειτουργούν ε, υπεύθυνα. Εάν λοιπόν ε, συμφωνήσει κανείς με, τον, ε, με τις ρυθμίσεις, τότε θα πρέπει να διορτηθεί κατά πόσον πρέπει να υπάρξουν και άλλες προϋποθέσεις. Η μελέτη, την οποία πρόσφατα κατέθεσε ο συνάδελφος κ. Φίτσι, δείχνει πόσα πολλά μέλη έχουν θεσπίσει τους σχετικούς κανονισμούς και κυρίως δείχνει ε, πώς ακριβώς διαφέρουν αυτά τα 18 καθεστώτα ε, και λόγω των ε, ε, το ότι πολλές φορές μιλάμε για συνεταιρισμούς και άλλες πάλι φορές μιλάμε για κεφαλοκικέ εταιρείε. Η διαφοροποίηση του δικαίου κατ' ουσίαν δεν αρκεί έτσι ώστε να αιτιολογηθεί η όλη λογική της κοινή αγοράς. Ε, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία ε, διασυνοριακή σημασία Βεβαίω οι περισσότεροι βασίζονται σε μετοχικές εταιρείε και τι περισσότερες φορές μόνο σε εισηγμένε εταιρείε, όπου αυτό το διασυνορικό στοιχείο είναι πολύ περισσότερο από ότι ε, σε συνεταιρισμούς οι οποίοι τις ε, περισσότερες φορές ε, ρυθμίζονται περιφερειακά. Όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας κανονισμός ευρύτερος, αλλά μπορεί κανείς να περιοριστεί σε εταιρείε όπου η διασυνοριακή δραστηριότητα είναι δυνατή. Σε πολλές μικρότερες επιχειρήσεις αυτό ε, δεν είναι απαραίτητο. Κατά την άποψή μου ε, θα έπρεπε να ρυθμίσει τα θέματα σε επίπεδο κράτους μέλους στο βαθμό ε, που δεν υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί. Μια ευρωπαϊκή ρύθμιση θα έπρεπε βέβαια να εστιασεί σε μεγαλύτερες ε, μορφές Δηλαδή να υπάρχουν εταιρείε που είναι συγμένες στο χρηματιστήριο ή είναι κεφαλογικές. Πέρα από αυτές τις αρμοδιότητες υπάρχει και η συνύπαρξη με υπάρχοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Παραδείγματο χάρη ο κανονισμός ε, για τα ευρωπαϊκά ταμεία ΟΕΣΕΦ. Επίσης ε, ε, και οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν στη χρηματοδότηση αλλά και στην υποχρέωση δημοσιοποίησης ορισμένων επιχειρήσεων. Ε, οι κοινωνικές επιχειρήσεις που εστιάζονται ε, στην κεφαλοχική αγορά, αυτό αφορά την ε, την επιθυμία της Κομισιόν και δεν ρωτάτε κανείς γιατί αυτή η πρωτοβουλία λείπει μέχρι τώρα. Κατά τα άλλα, το ερώτημα που αφορά στο επίπεδο ρύθμισης, αυτό το ερώτημα οδηγεί και στις ε, στη μορφή των ρυθμίσεων, επειδή οι νέες ευρωπαϊκές ε, μορφές όπως και η εναρμόνιση αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει να είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, εγώ θα ήθελα να προτείνω να παραμείνουμε στις υπάρχουσες μορφές, ε, δηλαδή στην, στις κεφαλοχικές εταιρείες. Και οι κοινωνικές επιχειρήσεις ε, μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε και το SE. Βεβαίω ε, δεν μπορεί κανείς ε, να γνωρίζει κατά πόσον αυτό το SE μπορεί να βασίζεται στο καταστατικό ή κατά πόσον πρόκειται μόνο για μια εξειδίκευση. Μια τέτοια εξειδίκευση θα μπορούσε να έχει διάφορες μορφές μεταξύ άλλων και τη μορφή μιας πιστοποίησης. Στο Αμερικανικό Δίκαιο υπάρχει παραδείγματος χάρη σε πάρα μια ειδική νομική μορφή, το Benefit Corporation. Από την άλλη υπάρχει πιστοποίηση B Corp, η οποία πιστοποίηση αποδίδεται από το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης B-Lab. Το γεγονός ότι όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις περνάνε μέσα από αυτήν την αμερικανική πιστοποίηση, αυτό το βρίσκω ε, θαυμάσιο ε, και ε, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα να μιλήσουμε για πραγματική ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Γιατί αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος να ισχύουν και στην Ευρώπη αμερικανικές προτεραιότητες Όπω όπως επίσης όπως συμβαίνει στο US IFRS. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η πιστοποίηση, αυτό σημαίνει ότι ε, όλα αυτά μπορούν να επεκταθούν περαιτέρω και στους ε, ευρωπαϊκούς ε, συνεταιρισμούς. Βέβαια, μια τέτοια πιστοποίηση αρκεί για να επιτύχουμε το να εκπέμψουμε ένα μήνυμα. Τώρα, το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρξουν υλικέ αλλαγές της νομικής βάσης ε, της ε, ε, ανώνυμης εταιρεία, αυτό εξαρτάται από το κατά πόσον αυτές οι εταιρικέ μορφές προσφέρουν στους μάνατζερ αρκετό περιθώριο για να πραγματοποιήσουν και αυτοί κάποιες σκέψεις για το κοινό καλό. Ε, παραδείγματο χάρη με ειδικέ επιτροπές και με την υποχρέωση δημοσιοποίησης. Λόγω της ειδική μορφής ε, της ανώνυμης εταιρεία, το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί γενικά, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή εδώ είναι απαραίτητο να υπάρξει μια νομική σύγκριση. Ε, τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Πρώτον, η πρωτοβουλία της Νομικής Επιτροπής έχει νόημα και είναι απολύτως απαραίτητη. Δεύτερον, προτεραιότητα θα έπρεπε να έχει η πιστοποίηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ ε, ένα καταστατικό χρειάζεται και προεργασία. Τρίτον, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στις εταιρικές επιχειρήσεις ε, ε, με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Εάν λοιπόν θα μπορούσα να προτείνω ο ευρωπαϊκός, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί να βασίζονται κυρίως σε κοινωνικές επιχειρήσεις ε, της κεφαλαίου ε, ίσως εντυρωτηθείτε ε, το κατά πόσον το να είναι εταιρεία εισηγμένη σε μία, στο χρηματιστήριο δεν έχει καμία σχέση με το να προσφέρει κοινωνικό έργο. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε όλο και περισσότερο για impact investment εδώ και ένα μήνα η πρώτη Benefit Corporation έχει εισαχθεί στην αγορά, αναφέρομαι στην Laureate Education, ε, εισήχθη ε, στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο και επιπλέον και σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν θέσεις ε, στο εμπόριο όπως Social Stock Exchange στο Λονδίνο ή Bolsa Social στη Μαδρίτη. Άρα δηλαδή αξίζει τον κόπο να συζητήσει κανείς για τη νομική βάση. Και χαίρομαι που αυτή τη ε, πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Να κλείσουμε αυτόν τον πρώτο γύρω νομικών προσεγγίσεων του θέματος και μετά παίρνουμε σε ερωτήσεις και απαντήσεις προς τους τρεις ομιλητές. Ο κύριος Μαρέκ Ιούχα, αντιπρόεδρος της κοινωνικής, του Επιμελητηρίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της Πράγας. Ε, έχετε κύριε 10 λεπτά το πολύ. Μετά από τις ε, δύο εισηγήσει ε, που άκουσα και μετά από αυτά που βιώνουμε στην Τσεχία, θέλω να σας πω ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο κανείς, όλοι μιλάνε γι' αυτό, αλλά κανείς δεν το έχει δει και κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί. όσον αφορά τώρα την ύπαρξή μας, υπάρχουμε εδώ και 8 χρόνια. Πριν από 8 χρόνια στο Σμιντήρν εγώ ως πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης και Εκπαίδευσης και ο συνάδελφός μου, ε, αρμόδιος για την περιφερειακή ανάπτυξη, διαπιστώσαμε ότι στην αγορά εργασίας ε, υπάρχουν ε, κάποια άτομα που δεν έχουν καμία προοπτική, διότι κατ' ουσίαν οι άνθρωποι αυτοί, αυτούς κανείς δεν θέλει να τους προσλάβει και να τους απασχολήσει. Εδώ και 27 χρόνια έχουμε εμπειρία στον τομέα αυτό και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον πολιτικό τομέα. Εδώ και 8 χρόνια είμαι δήμαρχος ε, σε μία μικρή περιοχή. Ο συνάδελφός μου απασχολείται στην ε, περιφερειακή κυβέρνηση και θα ήθελα να μου επιτρέψετε ξεκινώντας να σας παρουσιάσω ορισμένες βασικές αρχές. Δηλαδή, ε, τι σημαίνει κοινωνική επιχείρηση και ε, ποιον ακριβώς θα πρέπει να απασχολούν αυτές οι εταιρείες. Νομίζω ότι αυτό κανείς δεν το είπε. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ε, θα έπρεπε να μειώσουν την απασχόληση, θα έπρεπε να απασχολούν ε, πάνω από 40% ε, εργαζομένων με κοινωνικά κριτήρια. Έγινε επίσης λόγος για το κέρδος. Εμείς ε, συμφωνούμε ότι το κέρδος που απορρέπει την κοινωνία θα πρέπει να επανεπενδύεται και σε κοινωνικούς τομείς. Οι εταιρείε λοιπόν θα πρέπει να επιτρέπουν εξάλλου και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της επιχείρησης. Ποιοι είναι τώρα αυτές οι ομάδες στόχος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Είναι τα άτομα τα οποία έχουν ε, αναπηρία και είναι και επίσης οι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Δηλαδή ε, άτομα που αποκλείονται από το σχολείο, ε, προανφυλακισμένοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι. Αυτή είναι η ομάδα στόχος μας, η οποία πρέπει να προαχθεί στο, με τη μορφή των κοινωνικών επιχειρήσεων. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να γνωρίζει κανείς το εξή. Υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ε, κοινωνικές ε, υπηρεσίες, όπου προσφέρουμε υπηρεσίες ε, σε έναν πελάτη και ε, από κάτω αναφέρεται κοινωνικές επιχειρήσεις ε, που επιτρέπουν τον ε, προσπορισμό κέρδους. Ο πελάτης δεν είναι πια πελάτης, αλλά ένας συνεργάτης με σχέση εργασίας. Όλα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν κοινωνικές δυνατότητες. Η εταιρεία, επειδή είναι κοινωνική εταιρεία, πληρώνει φόρους και επίση η εταιρεία θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να προτιμάται, δηλαδή ε, να προσφέρει ε, κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν τον πελάτη να περάσει στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Ε, στον τομέα αυτό στην Τσεχία δεν υπάρχει νομοθεσία και επίσης εκταμείευονται κονδύλια και από τα κοινωνικά ταμεία. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί αυτών των ε, μειονεκτουσών ε, ομάδων. Ε, τώρα θα διερωτηθεί όταν μιλάμε για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τι σχέση έχουν αυτοί με τις ε, κοινωνικές εταιρείες. Δυστυχώς υπάρχει κάποια έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτούς που εκπονούν μελέτες και σε αυτούς που βρίσκονται κοντά στην πράξη. Ε, και όλα αυτά οδηγούν ε, στο να μην υπάρχει αποτελεσματική χρήση δημόσιων κονδυλίων. Πιστεύουμε ότι στην Τσεχία είναι πολύ καλή η κοινωνική στήριξη. Έχουμε τον νόμο περί απασχόλησης αναπήρων. Έχουμε επίση τα άτομα που υποφέρουν από κοινωνικό οικονομικό αποκλεισμό και αυτά μπορούν να απασχοληθούν από ενεργό πολιτική. Άρα δηλαδή και με τη βοήθεια του ε, Γραφείου εργασία μπορεί κανεί να στηρίξει ε, άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα. Πριν από λίγα χρόνια η τσεχική δημοκρατία αποφάσισε να μπορεί να αναθέτει έργο ε, σε ορισμένες ομάδες ε, με στόχο κατά κύριο λόγο το κοινωνικό στοιχείο ή ε, το να είναι ομάδες με αναπηρία. Πολλοί εργοδότες προτιμούν βέβαια τους χαμηλούς μισθούς αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ανοησία τουλάχιστον κάτω από, τα πρίσμα, από το πρίσμα που τα εξετάζουμε. Έχουμε περίπου 120 θέσεις απασχόλησης, τις οποίες δημιουργήσαμε για ε, μειονεκτούντα άτομα, αυτά που έχουν προβλήματα υγείας, ήταν 110, οι άλλοι είναι από άλλες ομάδες στόχο. Και διαπιστώσαμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι επιχειρήσεις με κοινωνική ένταξη, όπου οι εργοδότες ε, προέρχονται, έχουν σχέση με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι εργαζόμενοι εργάζονται για ένα χρονικό διάστημα, αποκτούν δεξιότητες και νομίζω εδώ θα πρέπει ε, να μπορεί κανείς να γνωρίσει και τα προσόντα του καθενός. Και το ερώτημα που τίθεται είναι... Ε, ποιο είναι το ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων. Μετά ακολουθεί η κοινωνική ενσωμάτωση, ε, δηλαδή η ενσωμάταση των μειονεκτούντων ε, εργαζομένων στην αγορά εργασίας και κατόπιν ακολουθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Που σημαίνει ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες επαγγελματικές δεξιότητες. Αναφέρομαι κυρίως σε άτομα με ε, κάποια αναπηρία ή κάποια καθυστέρηση. Βεβαίως ε, δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να αποκτήσει θέση απασχόλησης στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Αυτό που έχει σημασία είναι η εθνική νομοθεσία. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκτησει θεση απασχοληση στην περιοχή που βρίσκονται και πρέπει επίσης να είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα περίπου 20% του πληθυσμού που εμφανίζει αναπηρία. Αυτό το λένε οι μελέτες. Οι μελέτες είναι είτε με τη μορφή υγείας είτε κοινωνικής φύσεως. Ε, αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάσει και μέχρι το 40%. Ε, άτομα με ε, προβλήματα εκπαίδευσης, άτομα που θα αντικατασταθούν με ρομπότ. Ως εκ τούτου θα πρέπει να σκεφτούμε το ε, τι θα κάνουμε με τη χρηματοδότηση. Οφείλουμε ε, έξι μήνες νωρίτερα να ε, δηλώσουμε αυτές τις θέσεις απασχόλησης μέχρι να μας χορηγήσουν τα επιδόματα. Άρα δηλαδή εδώ οφείλουμε να προσφέρουμε δικό μας ίδιο κεφάλαιο. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ως προς τα εκπαιδευτικά συστήματα. Υπάρχει το θέμα της προοπτικής. Στους ε, μη κερδοσκοπικούς ε, οργανισμούς ε, εμείς προσφέρουμε την υπηρεσία, αλλά στην επιχείρηση ο εργαζόμενος εργάζεται για τον εργοδότη. Βεβαίω η δημόσια διοίκηση μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον ε, θα καταβάλλονται φόροι για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η δημόσια διοίκηση, η πολιτική, αυτοί θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα δίνουν τις παραγγελίες, θα αναθέτουν έργο σε τέτοιου είδους κοινωνικές επιχειρήσεις. Εγώ προσπάθησα να σας παρουσιάσω μια κυκλική δομή. Ε, στο κέντρο βλέπετε το πράσινο χρώμα, είναι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Το κίτρινο είναι το επιμελητήριο των κοινωνικών επιχειρήσεων και αυτό το μοβ χρώμα ε, είναι οι ενώσεις των εργοδοτών και όλα αρχίζουν από επάνω. Έχουμε τα άτομα με προβλήματα που εντάσσονται στην κάλυψη υπηρεσιών. Αυτό που λείπει εδώ είναι οι πελάτες να το κατανοήσουν ότι θα γίνουν εργαζόμενοι ε, σε μια κοινωνική επιχείρηση ή κάπου στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Δεν είναι πια πελάτες αλλά εργαζόμενοι και είναι σημαντική η ενσωμάτωσή τους. Για να λειτουργήσουν όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητο να ε, μεριμνά η δημόσια διοίκηση και να αναθέτει έργο αυτά, αυτές είναι οι επαφές μας, τα στοιχεία, μα, τα δικά μας. Βλέπετε τα τελευταία ε, τέσσερα χρόνια αποκτήσαμε πάνω από 40 μέλη και δημιουργήσαμε πάνω από 1.000 θέσεις απασχόλησης για άτομα με αναπηρία. Ερωτήσεις παρακαλώ από τους βουλευτές. Κύριε Ρέκνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένα τις εξή. Απευθύνομαι στον κύριο Φίτσε σχετικά με την προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί έχουμε κάνει και την εμπειρία μας με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ε, Πολλέ άλλε μορφέ απασχόληση και είδαμε ότι όλα αυτά δεν είναι απλά. Ε, δεν είμαι σίγουρη για το ποιο είναι το σημείο αναφοράς. Είπατε ε, μια προοπτική ε, SUP, μήπως μπορείτε λιγάκι να το αναλύσετε περισσότερο αυτό. Και κατόπιν, ε, ας δούμε λιγάκι τους ευρωπαϊκούς συνεταιρισμού. Κατά την τελευταία θητεία κάναμε την εμπειρία ότι παρότι θέλουμε τώρα όλα αυτά να τα εξυγχρονίσουμε, παρόλα αυτά η διασυνοριακή ε, προοπτική υποτίθεται δεν πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα από αυτού ε, και εμένα με ενδιαφέρει ε, να ξέρω πώς ακριβώς αντιμετωπίζετε εσείς την προστιθέμενη αξία. Προς τον καθηγητή κύριο Μέσλεν και προς εσάς μια ερώτηση. Αυτά που είπατε τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα για την πιστοποίηση. Ε, και λέτε ότι είναι πολύ δύσκολο να ε, συμπεριλάβει κανείς κάτι το καινούριο στο εταιρικό δίκαιο. Και εγώ θα ήθελα και επ' αυτού θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας το εξηγήσετε γιατί κάνατε κάποια ταξινόμηση ε, και μιλήσατε για έναν τέταρτο τομέα ε, θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο μιλήσαμε και ψηφίσαμε την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και αν τα συνδυάσουμε όλα τότε θα διαπιστώσουμε ότι ακόμα και εκείνων που ο στόχος τους είναι να προσποριστούν πολλά κέρδη, ακόμα και αυτοί κινούνται μέσα σε κάποια νομικά όρια και πρέπει να κινούνται μέσα σε αυτά. Άρα δηλαδή με την πρόταση την οποία καταθέσατε σχετικά με την πιστοποίηση δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι εντάξει αυτές είναι οι κανονικές επιχειρήσεις ε, είναι οι bad companies και μετά είναι οι άλλες επιχειρήσεις οι good companies. Μήπως θα πρέπει τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι όλες οι εταιρείε good companies, να εντάσσονται όλες ε, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να μην απαραίτητο να υπάρχει ένα πιστοποιητικό έτσι ώστε κάποιες που είναι καλές ε, να επιβραβεύονται με ένα είδος ε, πακέτου Marshall. Και τέλος, ε, μια ερώτηση προς τον κύριο Γιούχα, των ε, μηχανικών. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ε, βεβαίως θα πρέπει να έχουν μια τέτοια μορφή όπου θα πρέπει κανείς να έχει κατά νου ότι ο στόχος είναι να υλοποιηθούν κάποια στόχοι. Αλλά οι κυβερνήσεις, ή μάλλον με οι πολίτες, οι οποίοι κάποιοι εξ αυτών έχουν πολλά προσόντα, άλλοι όχι, πώς μπορούν όλοι αυτοί να αφομοιωθούν. Και πώς ακριβώς το φαντάζεστε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να τα κάνετε όλα αυτά ε, χωρίς ε, να ασκείτε ε, διακρίσεις. Γιατί αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη είναι ακριβώς αυτό. Πολύ συχνά είναι δύσκολο να συμπεριλάβει κανείς ε, κάποιους ε, επιτόπου, ίσως κάποιες μητέρες ή πατέρες ε, που δεν έχουν μεγάλη κινητικότητα και είναι αναγκασμένοι να προσέχουν τα παιδιά τους και τι συμβαίνει. Βρίσκεται κανείς κοντά στα σύνορα και από την άλλη πλευρά των σύνορων υπάρχουν εκείνοι που είναι πιο φτηνοί. Με άλλα λόγια, πώς μπορεί κανείς την κοινωνική επιχείρηση να την κρατήσει ζωντανή χωρίς να ασκεί και διακριτική μεταχείριση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου. Thank you very much. Uh, I will take all the... Λοιπόν, θα δώσω τον λόγο σε όλους, αλλά να είστε σύντομοι παρακαλώ. Δηλαδή ουσιαστικά είμαστε στο δεύτερο μέρος της ακρόασης, κύριος Μαστάλκα. Πρόεδρε, Ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίασή του, κύριε Πρόεδρε. και για την διοργάνωση αυτή τη τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση μαζί με την Επιτροπή Απασχόληση. Κάποιε ερωτήσει έχω. Αν κατάλαβα καλά, μα έλεγε ότι αυτέ οι επιχειρήσει πρέπει να έχουν σχέση με τι τοπικέ κοινότητε και αντίστοιχη υποστήριξη και δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλε, αν κατάλαβα καλά. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εναρμονισμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι δεν είναι, ερώτηση κάνω. Μπορούμε τότε να υπολογίσουμε τις επιπτώσεις, τις κοινωνικές και τις οικονομικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Ευχαριστώ. εκπρόσωπο τον κύριο Μπέκερ, ο οποίο δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Κύριο κύριος Μπέκερ μου ζήτησε να θέσω ορισμένα ερωτήματα στου εμπειρογνωμονε, Ποιος, ποια είναι η σχέση μεταξύ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των μελλοντικών εξελίξεων. Ποιο είναι το μέλλον της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τι είδου ε, επίσης δραστηριότητε διεκπαιρεώνουν καλύτερα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ποιες θα έπρεπε να είναι ιδανικά στα χέρια του δημοσίου των δημοσίων επιχειρήσεων Υπάρχουν άλλε επιλογέ εκτό από ένα νέο νομικό πλαίσιο για να βελτιώσουμε τι προοπτικέ των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ ωραία. Κύριος Λόπες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ερωτήσεις να κάνω μετά από τα ενδιαφέροντα που ακούσαμε από τους πυρογνώμονε. Καταρχάς, για τον αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν στις χώρες μέλη. 18 από ό,τι ακούσαμε. Οπότε αναρωτιέμαι, μπορούμε να υπολογίσουμε τον αντίκτυπο στις διάφορες νομοθεσίες για να αποφασίσουμε ποια θα πρέπει να προσαρμοστεί περισσότερο πανευρωπαϊκά. Υπάρχει κάποια έτσι διαφοροποίηση στις επιπτώσεις αυτών των νομοθεσιών ανάλογα με τη μορφή ή το καθεστώς της επιχείρησης. Βάσει τις εμπειρίες που έχουμε στις χώρες μέλη που είναι και επικύλη και πλούσια νομίζω έχουμε μια σοβαρή βάση δεδομένων σε σχέση με το τι είναι πιο αποτελεσματικό και τι προσφέρει περισσότερα κίνητρα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Καταρχάς αυτό. Δεύτερον, για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα που αφορούν και την Επιτροπή μας και που πρέπει να γνωμοδοτήσει αυτή την έκθεση. Υπόθηκε στην αρχή, αλλά λεπτομερώς μπορούμε να υπολογίσουμε τις επιπτώσεις της νομοθεσίας. Όχι μόνο τις ειδικές επιπτώσεις αυτών των επιχειρήσεων, που ξέρουμε, αλλά η νομοθεσία έχει άμεσο αντίκτυπο, ας πούμε, στην αγορά εργασίας, όπως, ας πούμε, άρση, εξάδεψη των διακρίσεων, κατανομή πλούτου, προσλήψης ατομών με αναπηρίες κλπ. Να ρωτήσω, λοιπόν, σχετικά χρειάζεται κάποια οδηγία για να το ρυθμίσουμε αυτό ή άλλα νομικά εργαλεία στην Ευρώπη. Και τέλος, ένα από αυτά που μας λένε όταν μιλάμε για συγκεκριμένη νομοθεσία στις αγοράς είναι οι στρεβλώσεις που διαφορετικές νομοθεσίες επιφέρουν στις αγορές. Εδώ ισχύει αυτό. Αυτά θέλω να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Κ. Ζανιέφ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν, καταρχάς μάλλον να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι, υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις αυτές είναι όλο και πιο δημοφιλείς. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, ένα νέο μοντέλο του επιχειρήν που δημιουργεί θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής του 2013, στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ε, δίνουν δουλειά σε πάνω από 14 εκατομμύρια ανθρώπους. Πιστεύω ότι πρόκειται για ανωδική τάση. Παρ' όλα αυτά, οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια. Έλλειψη αναγνώρισης, χρηματοδότησης, έλλειψη συνεκτικού νομικού πλαισίου. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερος ορισμός τους και περιχαράκωση του νομοθετικού πλαισίου. Έχει μεγάλη σημασία επίσης να αποσαφηνίσουμε το πλαίσιο λειτουργίας τους από νομοθετικής απόψεως και φως να τις διευκολύνουμε να αναπτυχθούν. Μία ερώτηση προς τον καθηγητή, τον κύριο Φίτσι. Μία από τις συστάσεις της μελέτης σας λέει ότι θα άξιζε έστω και μερικώς να εναρμονίσουμε τα πλαίσια λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Πιστεύετε ότι αυτό θα είχε πραγματικά ωφέλεια Κυρία Βερζιά. να είστε εκεί σύντομοι παρακαλώ. Γιατί... Α, γιατί μου το λέτε αυτό, επειδή είμαι η πρώτη γυναίκα που παρεμβαίνει και ξαφνικά μου λέτε να είμαι σύντομη. Ε, δεν το βρίσκω και τόσο κομψό, αλλά εν πάση περιπτώσει να συγχαρώ την Επιτροπή Γιώργη για την πρωτοβουλία της. Την περίμεναν πολύ Ο τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε και βάσει τη μελέτη νομίζω ότι είναι ιδανικός. Υπενθυμίζω ότι η Κομισιόν η ίδια όρισε την κοινωνική επιχείρηση στην Social Business Initiative την οποία όρισε ως ε, φορέα της οποίας ο βασικός στόχος είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος παρά το κέρδος. Αυτό αποτέλεσε και την κινητήρια δύναμη για την Κομισιόν. Πιστεύω το γεγονό μεταξύ άλλων ότι δημιουργήθηκαν τελευταία πάρα πολλέ θέσει εργασία από τι κοινωνικέ επιχειρήσει, οι οποίε ε, μάλιστα απέδειξαν και την αντοχή του στην κρίση, όπω υπογραμμίζει και η Επιτροπή. Το φαινόμενο άλλο παραμεληταίο είναι παρά ορισμένες αποτυχίες που πρέπει να αναλύσουμε. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια εναλλακτική πρόταση, κύριε Φίτση. Αξίζει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τη διαφορά αυτού που προτείνεται με αυτό που ισχύει σήμερα. Και θέλω να ρωτήσω το εξή. Προτιμάτε ένα γενικό πλαίσιο που αφήνει όμω ε, περιθώριο ευελιξία στις χώρε μέλη. Γιατί νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι η επικουρικότητα και η πρόθεση των κρατών να κρατήσουν πολλές αρμοδιότητες στα χέρια τους. Εμείς θέλουμε να καινοτομήσουμε στον τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω καλύτερα πώς θέλετε να προχωρήσουμε. Η σκέψη ήταν ενδιαφέρουσα. Εγώ θα ήμουν υπέρ τη δεύτερης εναλλακτική λύσης, ε, εάν πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ελπίζω η κυρία Σβερζιά θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η κυρία Ρέγκνερ είναι και αυτή η γυναίκα. Ευχαριστώ που συμφωνείτε μαζί μου. Το πρόβλημα είναι ότι είτε θα ζητήσουμε από τους προλαλήσεντες να απαντήσουν σε ένα λεπτό ή δεν ξέρω, ή πρέπει να κλείσουμε γρηγορότερα με τις ερωτήσεις. Διότι αλλιώς οι άλλοι δύο μιλητές πιστεύω ότι δεν θα έχουν καθόλου χρόνο να απαντήσουν και δεν μπορούμε να παρατείνουμε τη συνεδρίαση πέραν κάποιων λεπτών. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου λοιπόν με την προτινόμενη μέθοδο εργασία. Παρακαλώ. Ωραία. Κύριος Χουάν Αντώνιο Πεδρενοφρούτος, είστε πρόεδρος του Social Economy Europe. Έχετε τον λόγο για πόσα λεπτά. Δέκα λεπτά το πολύ. Θα σε λατρέψουμε αν, μας, αν σε 8 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχάς τη ευκαιρία που δείτε στο Social Economy Europe να μιλήσει εδώ σήμερα για την πρωτοβουλία εκπόνηση, ενός καθεστώτος κοινωνική επιχείρηση, επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας το οποίο θεωρούμε ότι πολύ σημαντικό για την κοινωνική οικονομία. Από το 2011, όταν θεσπίστηκε η έννοια της επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας, παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτής της πρωτοβουλίας, όπου ορίζουμε αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως παράγοντα κοινωνικής οικονομίας, όπως είπε η κυρία Βερζάτ. Επιχειρήσεις που σύμφωνα με αυτό τον ορισμό παρέχουν κοινωνικές επιχειρήσεις ή παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται σε ένα ευάλωτο κοινό λόγω ηλικία, μειονεκτήματος, αναπηρία κλπ. Προσπαθώντα να βοηθήσει την πρόσβαση στην αγορά εργασία των μειονεκτούντων ατόμων. Βάσει λοιπόν αυτή τη πρωτοβουλία, η Κομισιόν υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια διάφορα μέτρα που αποβλέπουν στην διευκόλυνση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Να ενισχύσει την παρουσία τους και να διευκολύνει το νομοθετικό πλαίσιο. Εμείς κάναμε διάφορες παρατηρήσεις σε σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Γιατί παρά τα θετικά που παρουσιάζει αυτή η πρωτοβουλία, έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα τμήμα της κοινωνικής οικονομίας. Με επιχειρήσεις που αφορούν την απασχόληση ή τις υπηρεσίες προς ευάλωτα άτομα. Αυτά ήταν, αυτές οι επιχειρήσεις ήταν το αντικείμενο της πρωτοβουλία της Κομισιόν, κάτι το οποίο περιορίζει το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας που είναι πολύ πιο ευρύ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πλειονότητα επιχειρήσεων, όπως οι συνεταιρισμοί, τα ιδρύματα, οι ενώσεις που έχουν οικονομική δραστηριότητα. Επιχειρήσεις κοινωνική πρόνοια επίση. και βεβαίως επιχειρήσεις κοινωνική επιχειρηματικότητας. Μιλάμε για όλα τα μεγέθη και όλου, όλων των ειδών επιχειρήσεις. Startups, μικρομεσαίε, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και που απαρτίζουν ένα μοντέλο επιχειρηματικότητα που εξυπηρετεί τον κόσμο. Και Όπω έλεγε ο καθηγητής Φίτσι, υπάρχει μια σύγχυση που ακόμα συνεχίζεται, γιατί υπάρχει σύγχυση μεταξύ των όρων κοινωνική επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχείρηση κλπ. Οπότε εδώ θα πρέπει να κάνουμε με διόρθωση ώστε να έχουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προωθήσουμε αυτό το είδος επιχειρήσεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε δύο πράγματα. Να έχουμε μια σαφή έννοια κοινωνική οικονομία που θα χρησιμοποιείται από όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και ιδιαίτερα από την Κομισιόν στις πρωτοβουλίε και στα μέτρα τα κοινωνικο-οικονομικά ώστε να μην περιοριζόμαστε μόνο σε ένα τμήμα σημαντικό τη κοινωνική επιχειρηματικότητα. Σημαντικό αλλά περιορισμένο όπω οι κοινωνικέ επιχειρήσει. Και δεύτερον θα πρέπει να αισθήσουμε από τις από τα θεσμικά όργανα μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που να εκμεταλλεύεται όλο το δυναμικό, το κοινωνικό-οικονομικό. Οι προτάσεις μας ως Social Economy Europe έγιναν δεκτές από την Κομισιόν και τα θεσμικά όργανα τα τελευταία χρόνια τέχθηκαν υπέρ της κοινωνικής οικονομίας. Το Κοινοβούλιο μέσω της, ε, της ομάδας του Intergroup για την κοινωνική οικονομία και αυτό ήταν ευήκο στα αιτήματά μας και εργάζεται συνεχώς υπέρ της κοινωνικής οικονομίας. Σε ένα ψήφισμα του Μάη του 2016 ζητείται από την Κομισιόν η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ώστε να απελευθερωθεί όλο το δυναμικό ώστε να έχουμε περιεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων. Το ίδιο και η ΟΚΕ σε έγγραφο που ζητά την εκπόνηση σειράς μέτρων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως τμήμα ενός μεγάλου και ευρέου προγράμματος για την προώθηση των αξιών της κοινωνικής οικονομίας. Και μάλιστα η ΕΟΚΕ τον Ιούλιο του 2016 ζήτησε από την Κομισιόν να περιλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της, εργασίας της το έγγραφο αυτό. Και οι χώρες μέλη παράλληλα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Οι τρεις τελευταίες ευρωπαϊκές διασκέψεις ζήτησαν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας σύμφωνα και ανάλογα με το βάρος της. Στο, στη δεύτερη, στο Λουξεμβούργο μάλιστα, υπό Λουξεμβουριανή Προεδρία, υιοθετήθηκε ένα έγγραφο που θα αποκαλούσαμε ιστορικό και που αναφέρει κοινωνική οικονομία ως σημείο κλειδί και κινητήρια δύναμη στην Ευρώπη. Και το Κοινοβούλιο ήδη είχε αναγνωρίσει στην ε, έκθεση του 2009 της Πατρίθια Τόγια της Ευρωβουλευτού το στοιχείο αυτό. Μάλιστα είχαμε και τη συγκρότηση μιας άτυπης ομάδας έξι κυβερνήσεων ήδη είναι 11 τα μέλη που παρακολουθούν ακριβώς την εξέλιξη της κοινωνικής οικονομίας και την ένταξή της στις πολιτικές τους. Και το Νοέμβρη στη Βλατισλάβα, το Νοέμβριο 16, υιοθετήθηκαν από 10 χώρες μέλη και υπεγράφησαν αυτά τα ψηφίσματα χώρες που ζητούν από την Κομισιόν οι πρωτοβουλίε για την κοινωνική επιχειρηματικότητα να υλοποιηθούν μέσω ενό Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράση για την κοινωνική οικονομία. Η Κομισιόν ανταποκρίθηκε και στην έκθεση εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται οι προτάσεις αυτές. Καταρχάς, η έκθεση τονίζει τη σημασία της κοινωνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Κοινωνική οικονομία και επιχειρήσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία. όπως είπε και ο κύριος Φίτση προηγουμένως. Ζητήθηκε επίσης από την Κομισιόν να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης. Και εμείς στο Social Economy Europe συμφωνούμε με αυτή την έκκληση γιατί χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική για το σύνολο της κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή για πάνω από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις και οντότητες της κοινωνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το 10% των επιχειρήσεων της Ένωσης που απασχολούν πάνω από 14 εκατομμύρια Ευρωπαίους, πάνω από το 10% της συνολικής απασχόλησης και που παράγουν το 8% της Ένωσης, οργανώσεις όπως ε, συνεταιριστικές, ιδρύματα, ενώσεις, επιχειρήσεις ένταξης, επιχειρήσεις κοινωνικής πρόνοιας προστασίας, ηθικές τράπεζες και οι κύριες οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας Βέλγιο, από Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Η Κομισιόν λοιπόν είχε ένα μόνιμο διάλογο μέσω του, της ομάδας του Intergroup και το κοινοβούλιο μέσω της ομάδας του Intergroup και η Διευθύντρια της Κομισιόν τη αντίστοιχη διεύθυνση για την κοινωνική οικονομία παρουσίασε πρόσφατα του έξι πυλώνε τη κοινωνική οικονομία που πρέπει να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια. Να ολοκληρώσω λέγοντα ότι για να συνεχίσουμε και να εδραιώσουμε αυτή την πολιτική πρέπει καταρχάς στην Ευρώπη να καθορίσουμε τα χαρακτηριστικά και να τα προσδιορίσουμε όπως αυτά που προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν κοινωνική οικονομία. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι κοινά που θα πρέπει να τηρεί κάποια επιχείρηση για να θεωρείται επιχείρηση κοινωνική οικονομία. Αυτό είναι βασικό και απαραίτητο για να χαραχτεί μια, οικονομία, μια πολιτική για την ανάπτυξη κοινωνική οικονομία στι χώρες μέλη. Προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα νομικό εργαλείο μη δεσμευτικό, συγκεκριμένα μια σύσταση που θα καθορίζει αυτά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής οικονομίας, ώστε κάθε χώρα μέλος, στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων, να ρυθμίζει τις επιχειρήσεις αυτές σύμφωνα με τις αξίες τους, τις βασικές, και να εντοπίσουμε τα μοντέλα επιχειρήσεων στην Ευρώπη που ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια και να τα προωθήσουμε. Έχουμε την χάρτα αρχών της κοινωνικής Οικονομίας που υιοθετήθηκε το 2002 υπάρχουν αυτά τα κριτήρια και είχαμε τι νομοθεσίες στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία κτλ. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μια κοινωνική οικονομία που να εξυπηρετεί τον κόσμο, του πολίτε. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό ο σκοπός, αλλά μέσο, ώστε να έχουμε απασχόληση ποιότητα, κατανομή πλούτου μεταξύ των απασχολουμένων στην επιχείρηση και γενικότερα στην κοινωνία για να βελτιώσουμε και τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων και των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή, μια μοντέλο μιας επιχείρησης αναπτυσσόμενης, βασιζόμενη στον κοινωνικό πυλώνα που θα συμβάλλει στην ποιοτική απασχόληση εντάσσοντας και περιλαμβάνοντας τους πιο αδύναμους ώστε να έχουμε μια πιο βιώσιμη οικονομία που δεν διευκολύνει την κοινωνική ένταξη, την τοπική ανάπτυξη και θα βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης. Εμείς στο Social Economy Europe είμαστε στη διάθεσή σας για να συμβάλλουμε στην έκθεσή σας ώστε να μετατραπεί αυτή σε στοιχείο πολιτικής για όλη την κοινωνική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φουτός. Ήσασταν πολύ πυκνός. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι είναι ενοχλητικό να μην έχει κανείς χρόνο και να πιέζεται. Και τώρα ο λόγος των καθηγητή Δόκτωρ Οκ Γιάννε. καθηγητή κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ντονάου στην Κρέμψη. Θα σας δώσω και εσάς 8-9 λεπτά για την παρουσίασή σας. Ο λόγος σε εσάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Σκεφτόμουν τι έπρεπε να πω, τι πρέπει να πω ως κοινωνιολόγος και ως ειδικό ε, στην κοινωνική καινοτομία. Είναι πολύ κοντά όλα αυτά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, στις κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Σκέφτηκα λοιπόν, να δούμε την επόμενη διαφάνεια, Παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Πολύ ωραία. Ελπίζω να μπορείτε να διαβάσετε τις διαφάνειες. Έλεγα λοιπόν... Um, how to consider how Σκέφτηκα λοιπόν να μιλήσω για το πώς η κοινωνική οικονομία συνδυάζεται με την κοινωνία. Δηλαδή πώς επικοινωνεί με συγκεκριμένους τομείς της κοινωνίας. Στην κοινωνιολογία από συστημικής απόψεως, από την απόψη των, της θεωρίας των κοινωνικών συστημάτων, θα λέγαμε ότι υπάρχουν τέσσερις ο νόμος, σταθερότητα και αλλαγή, που αποσκοπεί στο να επιτρέψει στους ανθρώπους να ζουν σε περιβάλλον δικαιοσύνης. Δεύτερον, η οικονομία, η οποία συμβάλλει στην κοινωνική ολοκλήρωση, την συνέχεια της κοινωνίας με τη διαρχή προσαρμογή στους διαθέσιμους πόρους, με συνεχή συγκερασμό αναγκών και πόρων, η ευμερία είναι το τρίτο, ε, ε, με συγχωρείτε η κουλτούρα, ο πολιτισμός είναι το τρίτο, το βλέπετε στη διαφάνεια, στο κάτω μέρος της οθόνης που ερμηνεύει τα νοήματα, το νόημα της ζωής, της ζωής με νόημα. Και ο τέταρτος τομέας είναι η πολιτική. Ο προσδιορισμός στόχων και η εξασφάλιση εν τέλει της ζωής σε ένα περιβάλλον ασφάλειας ασφάλεια στην εργασία, ασφάλεια κατά τη τρομοκρατίας, στην κοινωνική ασφάλιση και ούτω καθεξής. Μέσα σε αυτό το τετραμερές πλαίσιο λοιπόν διακρίνουμε αυτούς τους τέσσερις τομείς όπως είπα ο πρώτος τομέας είναι οι επιχειρήσεις, μετά έχουμε το δημόσιο, το κράτος, την κοινωνία των πολιτών, στη συνέχεια. Και εδώ, έχουμε, εδώ περιλαμβάνεται η κοινωνική οικονομία. Ο τομέας ο οποίος εργάζεται για το κέρδος είναι ένας συγκεκριμένος τομέας. Έχουμε τον μη κερδοσκοπικό τομέα. Οι επιχειρήσεις, ο κόσμος των επιχειρήσεων ζουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ο κοινωνικό τομέας όμως χαρακτηρίζεται από περισσότερη συνεργασία. Ο δημόσιο τομέα συγκεντρώνει στα χέρια του την ισχύ, την ισχύ την κρατική και βεβαίω την νομοθετική λειτουργία και την κανονιστική λειτουργία. Ενδιαμέσω θα δείτε στη διαφάνεια υπάρχουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι είναι οι ενδιάμεσοι διαμεσολαβητέ, αν θέλετε, οι οποίοι συμβάλλουν στην συνεργασία του πρώτου με τον δεύτερο τομέα συγκεράζουν τα κοινωνικά με τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία ονομάζουμε στην Αυστρία κοινωνική εταιρική σχέση. Δεν μπορώ να σας δείξω αυτό που θέλω, αλλά υπάρχει κάτι στη διαφάνεια που θέλω να τονίσω. Ευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο βασικών αυτών τομέων μέσω κάποιων ενδιαμέσων ο σχεδιασμό τη πολιτική γίνεται τριμερός. Έχουμε λοιπόν μια διονγκούμενη κοινωνική οικονομία η οποία συνδέεται τόσο με την ιδιωτική επιχειρηματικότητα όσο και με το δημόσιο, τους κρατικούς φορείς. Και η πρότασή μου προκειμένου είναι, αυτή είναι μια γενική σκέψη, είναι ότι η σε αυτή λειτουργία πρέπει να συμπεριλάβει εν τέλει τέσσερις διαφορετικούς εταίρους, τέσσερις διακριτούς εταίρους. Εσείς κύριε καθηγητά το ονομάσετε προηγουμένως ε, τέσσερις τομείς. Κάτι αντίστοιχο υποστηρίζω και εγώ εδώ. Πέραν αυτού, σκέφτηκα, τι είναι μια κοινωνική επιχείρηση. Έχει φυσικά κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε. Πρώτον, είναι μια επιχείρηση η οποία παράγει κέρδος. Δεν υπάρχει λόγος να τονίζουμε, δεν έχει νόημα να τονίζουμε την έλλειψη κέρδους. Το θέμα είναι, και εδώ είναι η διαφορά με τις άλλες επιχειρήσεις, πώς αξιοποιούνται αυτά τα κέρδη. Είναι κέρδη τα οποία επανεπενδύονται και προς τούτο πρέπει να υπάρχουν κέρδη για να μεγαλώσει η επιχείρηση και να αποφεληθούν και οι υπάλληλοι. Αυτό είναι το μοντέλο μιας καινοτόμου κοινωνικής επιχείρησης. Και το τρίτο, και ένα τρίτο μέρος αυτών των κερδών θα μπορούσε να επενδυθεί στην χρηματοδότηση κάποιων ε, κοινωνικών ε, ζητημάτων που υποστηρίζει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συγκεκριμένη συζήτηση. Όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να μπορούν να βασίζονται σε ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν είναι δυνατόν, υπεράνω των διαφορών από χώρα σε χώρα. Φυσικά, το μοντέλο πρέπει να προσαρμόζεται κατά τόπους. Ούτως ή άλλως έχουμε 18 διαφορετικές μορφές από ό,τι φαίνεται κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Χρειάζεται κρατόπους προσαρμογή. Το θέμα είναι η προσαρμογή αυτή να είναι πρώτον σύμβατη με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, τις πολιτικές για την εργασία κλπ. ώστε να δημιουργήσουμε ένα ούτως οικοσύστημα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Εν συνεχεία θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε στο πλαίσιο της κοινωνική ασφάλισης και κοινωνική πρόνοιας. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Μπέκερ. Έχουμε και τα κοινωνικά ζητήματα, όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Εκεί οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν ρόλο. Και δεύτερον, το θέμα είναι να καινοτομήσουμε πέραν των υφισταμένων μοντέλων, προσδίδοντας επιπλέον χαρακτηριστικά στο κοινωνικό μας μοντέλο. Ας πούμε, τεχνολογία. Πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Τι κάνουμε για την μεταβολή του κλίματος. Πώς ε, διαχειριζόμαστε την αλλαγή κλπ. κλπ. Οι κοινωνικέ λοιπόν επιχειρήσει μπορούν να τα συζητήσουν όλα αυτά με άλλες επιχειρήσεις, με τις κοινέ επιχειρήσεις, με το δημόσιο τομέα και με την κοινωνία των πολιτών, με ΜΚΟ και ούτω καθεξή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Δόκτωρα Χόκκιν, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε Είπατε επίσης ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ε, διωγγούμενο τομέα και ως εκ τούτου είναι σημαντικό για μας να έχουμε τέτοιου είδου συναντήσεις και σεμινάρια. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαστάλκα. Δύο λεπτά, μόνο δύο λεπτά όμως, για να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν χρειάζεται να μιλήσω. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να ακούσω απαντήσεις σε αυτά που ερωτήθηκαν. Χαίρομαι για τις απαντήσεις που θα δώσουν οι εμπειρογνώμονες. στο χρόνο που απομένει, αν έχει την καλοσύνη αγαπητοί προσκεκλημένοι, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας ετέθεσαν. Και δυστυχώς όμως ε, στις παρά 20 πρέπει να κλείσουμε. Κοιτάξτε, εγώ έχω το μόνο σας πω ότι δεν μπορώ να απαντήσω, ε, πρακτικά δύνατον. Και εδώ να κλείσω, να μην πω τίποτα άλλο. Αλλά η ευκαιρία το να υπάρχει αυτή η νομοθεσία είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τους νομοθέτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αναθέσει κάποιες ε, μελέτες που υπογραμμίζουν τη σημασία των κοινωνικών επιχειρήσεων ε, και των φορέων κοινωνικής μορφής στην Ευρώπη. Όλοι οι ευρωπαϊκοί ενωσιακοί θεσμοί έχουν ε, υπογραμμίσει σημασία αυτού του θέματος και έτσι εγώ αυτό το θεωρούσα δεδομένο. Η δική μου δουλειά ήταν να καταθέσω συστάσεις ε, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα καταστατικό κοινωνικό επιχειρήσεων. Αυτό το βρίσκω πολύ σημαντικό. Η όλη ιδέα του να έχουμε ένα ε, καταστατικό το οποίο θα σέβεται όλους τους πολιτισμούς στην Ευρώπη, αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό, κοιτάξτε η κοινωνική επιχείρηση ως ε, νομική οντότητα μπορεί να ικανοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες. Περισσότερο από άλλες απόψεις που λένε να έχουμε την κοινωνική επιχείρηση με μία συγκεκριμένη μορφή, με εταιρική μορφή. Τώρα από το πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά χρειαζόμαστε άλλη μία συνάντηση για να τα συζητήσουμε. Νομίζω όμως ότι στην έκθεση υπάρχει κάτι που μπορεί να αποτελεί τη βάση για μελλοντικές συζητήσεις. Άλλος από τους ομιλητές θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, θα απαντήσω τι ερωτήσει τη κυρία Ρέγκαν και του κυρίου Σούλτ ε, και τι δύο μαζί. Πρόκειται για την πιστοποίηση που θα ισχύουν για όλε τι επιχειρήσει σχετικά με την εταιρική ευθύνη. Ε, είναι αλήθεια ότι ο νομοθέτης επιβάλλει κοινωνιολογικές προϋποθέσεις σε όλους, αλλά και αυτό είναι περιορισμένο. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί ο νομοθέτης να επιβάλλει κάτι και αν το κάνει θα επιτύχει πολύ λίγα. Επειδή οι επιχειρήσει προφανώς και είναι προσανατολισμένε στο κέρδος, δεν μπορεί κανεί να ασκήσει υπερβολική πίεση. Ε, το πλεονέκτημα της πιστοποίηση είναι ότι μπορεί να απελευθερώσει δυνάμει της αγοράς, ότι ε, επιχειρήσει, αλλά και οι καταναλωτές ε, το επιβραβεύουν όταν επιχειρήσει συμπεριφέρονται με κοινωνικό τρόπο. Έχω λοιπόν κατά νου ένα είδος σήμανσης και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ε, μπορεί μια επιχείρηση να επιτύχει ε, καλύτερη θέση στην αγορά ε, και μπορεί να επιβληθεί στην αγορά ως good company. Άλλους παρακαλώ κανείς. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω ή μάλλον να πω, να προτείνω έναν ορισμό της ε, κοινωνικής επιχείρησης, ε, ορισμός τον οποίο χρησιμοποιώ εγώ, ε, πρόκειται για μια υπεύθυνη μεταχείριση ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά. Και με βάση αυτό θα πρέπει κανείς να ορίσει πώς είναι δυνατόν να προαχθούν όλες αυτές οι ομάδες γιατί χωρίς την ε, περιφερειακή ε, προαγωγή, την πρόθεση από τις εθνικές ε, κυβερνήσεις που γνωρίζουν πολύ καλά τι είδου προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες, αυτοί όλοι θα πρέπει να τα ορίσουν γιατί οι επιπτώσεις και η επαρρύθμιση των επιπτώσεων είναι αυτά που έχω πει. Είτε δηλαδή θα πληρώνουμε με τα χρήματα των φορολογουμένων τις ε, κοινωνικές παροχές, είτε θα αφήνουμε στις επιχειρήσεις περιθώριο ε, για επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλα σχόλια. Κατόπιν τούτου ευχαριστώ όλους ε, τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και επίσης να ευχαριστήσω ε, και τη συμπρόεδρο που με βοήθησε το σημείο υπερθμών 18 του κυρίου Μαστάλκα που δεν το εξετάσαμε σήμερα. Θα το εξετάσουμε αύριο μετά τις ε, ψηφοφορίες. Γεια σας.